στην ημερήσια διάταξη, θα πρέπει να καθορίσουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα και για αύριο. Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης που έχει οθετηθεί από, τους, από τη των Προέδρων στις 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το άρθρο 130, έχει διανεμηθεί και μετά από διαβουλεύσεις πολλές με τις πολιτικές ομάδες, προτάθηκε και συμφωνήθηκε να γίνουν οι κάτωθοι αλλαγές. Τετάρτη, σήμερα, 23 Μαρτίου του 2011, συζήτηση για τη δήλωση Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση στην Ιαπωνία είναι ένα σημείο που θα προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη, καθώ και το θέμα των ε, συναγερμών για, την, ε, για τα προβλήματα των πυρηνικών αντιδραστήρων. Θα αντικαταστήσει τι δηλώσει ε, του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γυτνίαση που αναβάλλεται για τον Απρίλιο, δηλαδή σε 15 μέρε. Έχει υποβληθεί σχετικό κείμενο και θα ψηφιστεί την Πέμπτη για την Ιαπωνία. Δεύτερο. Δεύτερη αλλαγή. Έκθεση Μπαλζάνη για την προετοιμασία για το κατάρτιση προπολογισμού 2012 θα συζητηθεί την Πέμπτη σαν δεύτερο σημείο μετά την κοινή συζήτηση για τις συμφωνίες για τις αερομεταφορές. Τρίτη αλλαγή, την Τετάρτη, για την Τετάρτη πάντα, προφορική ερώτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων συμπεριλαμβανομένης και τιμής για ε, το πετρέλαιο από σχιστόλιθο και από την άμμο. Ε, δεν θα υπάρξει ψήφισμα. Τέλος, τέταρτη αλλαγή που αφορά την Τετάρτη έκθεση του συναδέλφου του κυρίου Τσίτσεστερ όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και την Υπηρεσία για την Ασφάλεια. ευρωπαϊκό Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Αυτό άνευ συζητήσεως θα συμπεριληφθεί στο χρόνο ψηφοφοριών για την Πέμπτη. Και τώρα αλλαγές όσον αφορά το πρόγραμμα της Πέμπτης, αύριο δηλαδή 24 Μαρτίου. Πρώτα απ' όλα έχουμε την έκθεση Simpson Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, αναβάλλεται αυτό το θέμα για την Σύνοδο του Απριλίου. Δεύτερη αλλαγή, έκθεση Μορέιρα για περαιτέρω μακροοικονομική βοήθεια για τη Γεωργία και αυτή αναβάλλεται για την Σύνοδο του Απριλίου. Και τέλος, η ψηφοφορία για πρόταση ψηφίσματος για αλευτική συμφωνία Μαυριτανίας, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ενώσεως αναβάλλεται για μία από τις μελλοντικέ μας συνόδους της Ολομέλειας. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι αλλαγές που συζητήθηκαν με τις πολιτικές ομάδες και οι πολιτικές ομάδες εξέφρασαν σύμφωνη γνώμη. Αυτό σημαίνει ότι η ημερήσια διάταξή μας έχει καταρτιστεί και προχωράμε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Η έκθεση του κυρίου Μπροκ και του κυρίου Γκουαλτιέρη σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη-μέλη με νόμισμα το ευρώ.